Το επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Δανέλη για την γαλάζια ανάπτυξη, πρόωθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού. Πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Βασική αιτία της μεγαλύτερης κρίσης χρέους που έχει γνωρίσει η Ένωση καθώς και της συνακόλουθης κοινωνικής μάστιγας της ανεργίας που με εφιαλτικούς ρυθμούς συνεχώς διευρύνεται είναι το ότι η ευρώπη έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της. η ανάδυση νέων παγκόσμιων παιχτών την εκτόπισαν από τις πρωτοπορίες της παγκόσμιας οικονομίας. πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως να στραφεί σε νέα αναπτυξιακά πεδία. η στροφή στη θαλάσσια οικονομία και τους πλουτοπαραγωγικούς θαλάσσιους πόρους αποτελεί μια φιλόδοξη οραματική αλλά ταυτόχρόνω ρεαλιστική πρόταση ανοίγει προοπτικές για ευρείες συνεργασίες μεταξύ οικονομικών κλάδων που δεν δραστηριοποιούνται μονάχα στις παράκτιες περιοχές της ένωσης των 28 πλέον από σήμερα χωρών μελών αλλά στο σύνολο της επικράτειάς της. Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός σε όλες τις θεματικές του εκφράσεις, η υδατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η θαλάσσια εξόριξη ορυκτών, καθώς και μέσω αυτών η ενίσχυση της ναυτιλίας και της χυμαζόμενης ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελούν τους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης που μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος της θαλάσσιας οικονομίας σε 590 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 και με κατάλληλες πολιτικές κατάρτισης που να εξασφαλίζουν ένα ευκίνητο εργατικό δυναμικό με επαρκή εξειδίκευση και εμπειρία η συνολική απασχόληση στη γαλάζια ανάπτυξη δύναται να ξεπεράσει την εκτίμηση των 7 εκατομμυρίων θέσεων εργασία μέχρι το. 2020. οι τοπικέ περιφερειακέ εθνικέ και ευρωπαϊκέ αρχέ θα πρέπει να δημιουργήσουν τι απαραίτητε προποθέσει για βιώσιμη ανάπτυξη όπω συστήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών αναβάθμιση των υποδομών πρόσβαση σε επαγγελματικέ δεξιότητε διάχυση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και βεβαίω εξασφάλιση επαρκού χρηματοδότηση. προκειμένου οι τομεί τη γαλάζια ανάπτυξη να εξελιχθούν και να ξεδιπλώσουν το σύνολο τη δυναμική συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι αναγκαίο ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο ευρωπαϊκή ένωση σε ό,τι αφορά το συντονισμό και τι συνεργασίε μεταξύ των υφιστάμενων πολιτικών καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλειών και εργαλείων. βεβαίως για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η γαλάζια ανάπτυξη οι φορείς δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να εργαστούν σε ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη του τις νέες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης. σε μια εποχή περικοπής δημοσίων επενδύσεων στα κράτη μέλη είναι επιτακτική ανάγκη οι αναπτυξιακές πολιτικές και κυρίως τα έργα υψηλού κόστους όπως είναι αυτά των μεταφορών των επικοινωνιακών και ενεργειακών υποδομών να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου είκοσι, αλλά βεβαίως και μετά από αυτήν. Είναι ανάγκη να διοχετευτούν οι διαθέσιμοι πόροι των Ευρωπαϊκών Ταμείων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών σε έργα της γαλάζιας οικονομίας τα οποία είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν σε προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. πρωταρχική προϋπόθεση και βασική πρόκληση αποτελεί η διασφάλιση της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας της γαλάζιας ανάπτυξης ότι δηλαδή δεν θα βλάψει το ιδιαιτέρως ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμβάλει παράλληλα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. οι λαοί της ευρώπης τα τελευταία 9.000 χρόνια στρέφονταν οργανωμένα στη θάλασσα αναζητώντας και διασφαλίζοντας καλύτερο μέλλον. Κυρία Επίτροπε, χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση τη Επιτροπή για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και ζητούμε την επίσπευση των διαδικασιών και την ανάληψη από μέρου σα κάθε πρωτοβουλία που είναι αναγκαία για τη στήριξή τη. Τέλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά όλου του κοιόδη εισηγητέ για την εξαιρετική συνεργασία μαζί του, καθώς και όσου εργάστηκαν για την τελική διαμόρφωση της έκθεσής μα. Σα ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ τους ομιλητές. Κυρία Πατράου Νάβες πρώτη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή, τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή για τη συμβολή τους στην ε, ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης, πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης για τις θαλάσσιες ε, περιοχές, τις παράκτιες, για την αυπηγική, την έρευνα, την καινοτομία, την εξόριξη ε, από το θαλάσσιο βυθό. Και η σκιώδης ε, έκθεση ε, σημειώνει ότι δεν έχουμε αρκετά ε, προχωρημένη τεχνολογία για την εξόριξη από το θαλάσσιο βυθό. Πρέπει να γίνουν μελέτες σκοπιμότητας προκειμένου να δοθεί επαρκής ενημέρωση, νομιμοποίηση εντό εισαγωγικών για αυτή την εξόριξη με ε, τεχνολογία που θα επιτρέπει και βιωσιμότητα βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με 2 εκατομμύρια ευρώ το έργο μήτας ε, για να συλλέγονται στέρεα δεδομένα για την εξόριξη του θαλάσσιου βυθό Πρέπει να αξιοποιούμε τους, τον πλούτο βεβαίως ε, του πλανήτη, αλλά αυτό κατά τρόπον αηφόρο, κατά τρόπον οικολογικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συγχαίρω τον εισηγητή για αυτή τη λεπτομερή έκθεση του που όντως συνδυάζει τις διάφορες πολιτικές, τι τομεακές για την ε, θαλάσσια πολιτική. Δεν μπορεί να υπάρξει γαλάζια ανάπτυξη αν δεν υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική νοοτροπία που έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Εδώ μιλούμε για πάρα, πολλά, πάρα πολλές ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όλα τα θεσμικά όργανα. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία ασχολούνται με θέματα ε, θαλάσσιας πολιτικής ή ναυτικές σχολές, οι οποίες δεν είναι τελικά πολύ δημοφιλείς. Επίσης η καριέρα, η ε, ε σε αυτόν τον κλάδο δεν ευδοκιμεί. Οι χώρες λοιπόν που είναι θαλάσσιες θα πρέπει να έχουν σαφείς στρατηγικές και ολοκληρωμένες πολιτικές σχετικά με την την ε, εκμετάλλευση των θαλασσίων πόρων. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρξει και ένα ε, εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ε, μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αναφέρω ότι πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα της ανάπτυξης της στρατηγικής για την Μαύρη Θάλασσα, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι το 2020 θα έχουμε πάρα πολύ ε, αυξημένο πληθυσμό στην, ε, ε, στη γη. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένε πολιτικές πια. Η Ευρώπη έχει ένα αρκετά μακροπρόθεσμο όραμα και έχει εκπονήσει τις σωστέ πολιτικές, αλλά πάντα υπάρχουν πάρα πολλέ πολιτικέ οι οποίες χρειάζονται περισσότερη έρευνα σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια πολιτική. Πρέπει λοιπόν την έρευνα να την χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερα έτσι ώστε να έχουμε πιο βιώσιμη πολιτική για τη θάλασσα. Μιλούμε για την ε, γαλάζια ε, ανάπτυξη και η οποία βεβαίως είναι κομμάτι τη ε, στρατηγικής για το 2020, για την ανάπτυξη και για τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να αναπτύξουμε την γαλάζια βιοτεχνολογία που, είναι, που μιλούμε για τη χρήση της μόνο σε ένα επίπεδο 10%, μιλούμε για α, ορυκτά πρώτες ύλες. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι θέλουν να, ε, να τρώνε όλο και περισσότερα ψάρια. Πρέπει λοιπόν τα αποθέματα που υπάρχουν να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ευχαριστώ και την Επίτροπο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ. Ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλουμε πράγματι να αναπτυχθεί η γαλάζια οικονομία, αλλά αυτή πρέπει να είναι και πιο πράσινη. Γιατί σίγουρα πολλά επαγγέλματα εξαρτιόνται από τη θάλασσα, αλλά και πολλές φορές έχουμε και ρήπανση του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Θέλουμε λοιπόν μια οικονομία γαλάζια που θα ενισχύσει και θα αυξήσει τις δραστηριότητες γύρω από το θαλάσσιο ε, πλούτο αλλά διατηρώντας μακροχρόνια αυτόν τον πλούτο να βοηθήσει στην κοινωνική συνοχή και σε νέα επαγγέλματα που πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν σπουδάσει αλλά δεν βρίσκουν εφαρμογές ε, στις σημερινές πολιτικές. θέλουμε επίσης ε, σωστά σχέδια θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης έτσι ώστε πράγματι η γαλάζια οικονομία να αποβεί προς όφελος και του περιβάλλοντος και της απασχόλησης και της οικονομίας. Ευχαριστώ. Μοργάντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται από μια περιοχή την Τοσκάνη που έχει έφεση ναυτιλιακή και γνωρίζει λοιπόν τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες του, του κλάδου. Θα πρέπει να αναφερθώ στα πρόβλημα που, προβλήματα που προκύπτουν από την οδηγία περιπηρεσιών που πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι συμβάλλουν στην ευημερία και την ασφάλεια των ε, ναυτιλιακών μεταφορών. Ε, Εμεί στην Ιταλία γνωρίζουμε την ε, φιλοξενία και την σημασία που έχει ο κλάδος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε λοιπόν να επηρεαστεί από άτομα άσχετα τα οποία ασχολούνται με τον κλάδο, διότι όσοι ασχολούνται με τον κλάδο αυτόν, όπως εγώ, το γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχουν μειονεκτικές περιοχές, νησιωτικές κλπ. Η δημιουργία ελεύθερων ζωνών θα μπορούσε να είναι κάτι το χρήσιμο, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί άνετα και αποτελεσματικά στην ίσο Έλμπα, που τα τελευταία χρόνια γνώρισε ύφεση και θα μπορούσε λοιπόν να ενισχυθεί με διάφορες φορολογικές διευκολύνσεις και επενδύσεις. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Εσάιερ. Πρόεδρε, η Ιρλανδική Προεδρία που μόλις ε, ολοκληρώθηκε ασχολήθηκε με το θέμα της ε, γαλάζιας ανάπτυξης ε, και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στον τομέα αυτό πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας υπήρξαν πάρα πολλά δύσκολα ζητήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν αλλά έχουμε τελικά αυτή την πολύ καλή γνωμοδότηση πια και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί τονίζεται όντως η γαλάζια ανάπτυξη. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω μόνο για την υδατοκαλλιέργεια και για την αλληλεία, αυτά τα συζητούμε πάντα, αλλά και για τη γαλάζια ενέργεια για, την χρήση ε, των ε, μεγάλων ε, για τις ανεμογεννήτριες. Στην Ευρώπη βεβαίως δεν έχουν πάρα πολλά κράτη τις ε, κατάλληλες δυνατότητες, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα να γίνει αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να, κάνουμε, να λάβουμε υπόψη μας και τα όσα προβλέπει ο ΠΟΕ. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή και να υπογραμμίσω δύο θέματα τα οποία θεωρώ πως ε, χρήζουν ιδιαίτερη σημασία ε, το πρώτο ζήτημα για μια ανάπτυξη αηφόρου και ισορροπημένη <clears throat> είναι να δημιουργήσουμε ολοκλήρωση ανάμεσα στην στις ακτές και την υπηρετική χώρα. <clears throat> Υπάρχει μια βουλημική λογική που καταπατάει τις, τους πολιτισμούς και τις αξίες ε, ενώ υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες ε, θα μπορούσαν να εποφεληθούν και να δημιουργήσουν έτσι κίνητρα για τους ε, ε, κατοίκους της περιοχής. Θα ήθελα να πω ότι θα είμαστε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το θέμα της υδαροκαλλιέργειας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στην υδαροκαλλιέργεια η χρησιμοποίηση αντιβιωτικών και κάποιων τροφών δημιουργεί ανισορροπία στο οικοσύστημα και δημιουργεί επίσης ευτροφισμό από προϊόντα τα οποία περιέχουν φόσφορο και νάτριο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Επίτροπος τώρα θα πάρει το λόγο για να ολοκληρωθεί και ο κατάλογος των ομιλητών. Thank you, President. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Δανέλη, τον εισηγητή, καθώς και τους σκιώδησίτες, αλλά και τα μέλη των Συνομωδίων επιτροπών. Είναι Επιτροπή Μεταφορών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και βεβαίως Αλίας. Κατήρτισαν ένα εξαιρετικό κείμενο και χαίρομαι που όλοι οι ομιλητές χωρίς καμία εξαίρεση αναγνώρισαν ότι στην έκθεση και στην έκθεσή μας για την γαλαζία ανάπτυξη. Διατυπώνονται μακρόπνες προοδευτικές προτάσεις σε ένα αυτοσυνεπές πλαίσιο. Χαίρομαι επίσης διότι η έκθεση υπογραμμίζει τους πέντε τομείς που τονίζει και η Κομισιόν, που είναι και οι τομείς στους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να κοινοτομήσουμε. Αυτοί οι πέντε τομείς είναι η γαλαζιανέργεια, οι ηχθειοκαλλιέργειες, ο παρακτήριος η οι εξορίξεις, εξορίξεις και η βιοτεχνολογία. Επιτρέψτε μου να πω και τα εξή πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, όσον αφορά την ναυτιλία, τι θαλάσσιε μεταφορέ και την ναυπηγική. Όντω, αντιμετωπίζουμε δυσκολίε, όπω άλλωστε υπογράμμισαν ο εισηγητή και άλλοι μιλητέ. Όμω, θα ήθελα να υπογραμμίσω επίση ότι μπορούμε με πολλού διαφορετικού τρόπου να τονώσουμε την βιώσιμη αναπτύξη τομέα, Μειώνοντα τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, εξελίφοντα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και προωθώντα την καινοτομία. Υπάρχει λοιπόν ακόμη και εδώ περιθώριο βελτίωση όσον αφορά τον παράκτιο τουρισμό. Συμφωνώ με την έκθεση. Η βασική πρόκληση, προκειμένου, είναι να διασφαλίσουμε ότι θα εξεύρουμε το απαραίτητο εργατικό δυναμικό με τις σωστές δεξιότητες. Και αυτό το πετυχαίνουμε με την ανακοίνωση της Επιτροπής που θα εκδοθεί πριν από τα τέλη του 2013. Τέλος, όσον αφορά την σημασία της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες ορισμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη εξασφάλισης αηφορίας σε όλες αυτές τις δράσεις. Συμφωνώ ότι η περιβαλλοντική διάσταση πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε πρωτοβουλία στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης. Οφείλουμε να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, εάν βεβαίως θέλουμε να υποφεληθούμε και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει και όχι να το καταστρέψουμε όπως κάναμε σε μερικές περιπτώσεις στο παρελθόν. Γι' αυτόν τον λόγο, της εξόρυξης σε θαλάσσιες περιοχές και το θέμα των περιοριστικών επιπτώσεων ε, είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο και το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα για, την, για τις εξορίξεις επαναλαμβάνω είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει καμία εμφολία. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας στην ανακύκλωση. Όμως ακόμη και έτσι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εξασφαλίσουμε σταθερή ροή των υλών που χρειάζεται βιομηχανία. Η πρότασή μας λοιπόν είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις. Οι εξορίξεις στη θάλασσα θα δημιουργήσουν αίσθηση θέσεις εργασίας, άλλες ευκαιρίες, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά και θα εξασφαλίσουν εγγυήσει για την προμήθεια πρώτων υλών. Βεβαίω με προποθέσει. Και εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή και άλλου ομιλητέ. Υπάρχει ένα προαπαιτούμενο. Αυτό ο νέο κοινοφανή Τομέα, αλλά αυτό ισχύει και για κάθε άλλο τομέα, πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αηφορία. Με άλλα λόγια και πιο συγκεκριμένα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εάν κάποιο εργαλείο του ανθρώπου αγγίξει τον πυθμένα της θάλασσα, πρέπει αυτό να γίνει με πλήρη σεβασμό περιβαλλοντικών κριτηρίων. Και αυτό θα πράξουμε. Και έτσι θα γίνει. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους ομιλητές καθώς και όλους τους βουλευτές για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας για την γαλάζια ανάπτυξη. Εγώ ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας της διάταξης. Έκθεση της κυρίας Τόια, συμβολή των συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση της κρίσης. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε.